Θα έλεγα να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίαση. Θα προεδρεύσω σήμερα, διότι η πρόεδρός μας βρίσκεται σε ένα τριμερή διάλογο σήμερα το απόγευμα. Οπότε θα αναλάβω τα καθήκοντά της. Θα προσπαθήσω να σας διασκεδάσω σήμερα το απόγευμα. Εδώ ε, νομίζω για, την, ε, για τον κανονισμό της κοινής αγοράς ε, μετά από αίτηση των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών αναβάλλεται επειδή και οι υπόλοιποι συμφώνησαν. Το σημείο λοιπόν 7 ε, από την ημερήσια διάταξη αναβάλλεται για το σχέδιο ημερήσιας διάταξης Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται και περνάμε στις ανακοινώσεις. Να καλωσορίσω όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, web streaming. Άλλωστε είμαστε και η υπεύθυνη επιτροπή για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Και για την εφαρμογή meeting ξέρετε ότι διατίθεται σε όλους τους ε, βουλευτές την ε, στους βοηθούς και σε όλους τους συνεργάτες μας. Στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 4ης Ιουνίου. Ε, τα πρακτικά, ε, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Εγκρίνονται λοιπόν, οπότε προχωρούμε στην ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους και τις εκδηλώσεις. Πρώτο σημείο είναι η ομάδα εργασίας στην οποία προεδρεύω εγώ για την πνευματική ιδιοκτησία και την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συναντηθήκαμε στις 23 Ιουνίου για το θέμα αυτό. Ασχοληθήκαμε με τον τομέα των οπτικοακουστικών και αυτό που προέκυψε με τις παρουσιάσεις από τους δημιουργούς και τους ε, καλλιτέχνες από ενώσεις καταναλωτών και πανεπιστημιακούς. Είχαμε μια τόσο πολύ, μεγάλη πολυφωνία για την περιπλοκότητα του ζητήματος αυτού που ξέρουμε ότι εγγύζει πολλούς διαφορετικούς τομείς εντός των οποίων ούτως ή άλλως υπάρχει μεγάλη περιπλοκότητα. Έμαθα πολλά λοιπόν για το πώς χρηματοδοτείται ο τομέας, η κινηματογραφική βιομηχανία, η δημιουργή, ή σεναριογράφοι, των ταινιών, αλλά υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιληθούν και από άποψη πανεπιστημιακή υπάρχουν ακόμη διαφορετικές απόψεις, αντικρώμενα επίσης συμφέροντα. Οπότε είναι πολλά αυτά που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Και ίσως η Τζούλια που είναι και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων Ε, θα μας επιβεβαιώσει αν η πρώτη πρόταση για τα πνευματικά δικαιώματα δεν πρόκειται να έρθει έτσι καλώς πριν από το χρόνο το Γενάρη γιατί χρειάζεται όλη αυτή η περισυλλογή προηγουμένως. Και μπορεί και να καθυστερήσει. Και καλό είναι τα πάντα να τα έχουμε μελετήσει σωστά πρέπει να γίνει μια βιαστική πρόταση. Πάντω, η ομάδα εργασία θα συνεχίσει τι εργασίε τη. Η επόμενη συνεδρίαση είναι την Πέμπτη το πρωί. Και ένα συνάδελφο ω αναπληρωτή θα παραστεί ω εκπρόσωπό μα. Είναι σημαντικό η Επιτροπή μα να είναι δραστήρια και ενεργή. Υπάρχουν ήδη σχόλια και αντιδράσει και αυτό είναι ένα σημαντικό έργο τη δουλειά μα. Υπάρχουν σχόλια από του συναδέλφου. Τζούλια, θε να προσθέσει κάτι. Just uh, Απλώς να προσθέσω ότι στη συνεδρίαση της Πέμπτης το πρωί θα μιλήσουμε για την, για την ελευθερία έκφρασης ε, και θα παραστώ ως ε, μέλος και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Νομίζω ότι αυτό ήταν σημαντικό να τονιστεί και δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της Επιτροπής. Το πρωί μόλις με ενημέρασαν για το χρονοδιάγραμμα του Ιανουαρίου, αλλά περιμένουμε περισσότερε εξηγήσει από την Επιτροπή. Ξέρω ότι θα έχουμε ένα πληρωτή από κάθε ε, πολιτική ομάδα, θα υπάρχει ποσοτική εκπροσώπηση. Ο Νταν θα μας Ε, ε, ενημερώσει, αλλά επειδή το πανόραμα είναι ένα σημαντικότατο θέμα, θα το δούμε. Ε, την Πέμπτη εγώ δεν θα μπορέσω να παραστώ γιατί πρέπει να είμαι και πάλι στη Σκοτία για μια συνάντηση στη Γλασκόβη. Αλλά δεν φταίω εγώ γιατί συνάντηση αρχικά είχε προγραμματιστεί για Τετάρτη. Εάν οι συνάδελφοι συμφωνούν μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Θα μιλήσουμε εδώ λοιπόν για το θέμα των για τα προϊόντα φωκών. Ο κύριος ε, Σουάπ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω ότι ο συνάδελφος που είναι αρμόδιος στο θέμα αυτό δεν μπόρεσε να παραβλεφθεί σήμερα, γι' αυτό μας μου ζήτησε να σας παρουσιάσω τι έγινε στον τρομερή διάλογο την προηγούμενη Πέμπτη. Και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Μου είπε λοιπόν ότι ήθελε να μα ενημερώσει. Ότι την προηγούμενη Πέμπτη, όταν έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος, και ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσει. Είναι μικρό το θέμα αυτό και γι' αυτό λοιπόν κατάφεραμε του συναδέλφου να ολοκληρώσει σε αυτή την πρώτη συνάντηση τις διαπραγματεύσεις. Είναι αισιόδοξο ότι θα είναι καλέ ειδήσει από πλευρά του Συμβουλίου μετά την κοροπέ της Γιατί πρόκειται μόνο για μεταφορά απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού εργασία, την οποία και επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία που συνάδει με τον κανονισμό του ΠΟΕ και ε, καταργεί τις εξαιρέσεις MRM, αλλά κρατά την εξαίρεση για τους Ινουίτες. Και σύμφωνα λοιπόν με τη διαταξή αυτή, τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τις κοινότητες των Ινουιτών μπορούν να διατίθενται στην αγορά γιατί λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των κοινοτήτων αυτών. Το είχαμε συζητήσει το 2008 το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο. Το θέμα δεν είναι οι καθημερινές ε, δραστηριότητες των Ινουητών, αλλά κυρίως η εμπορία των προϊόντων αυτών από την θύρευση φώκιας. Η απόφαση λοιπόν την οποία ελπίζουμε θα επιβεβαίωσει το Συμβούλιο αύριο θα επιτρέψει αυτά που έχουμε αποφασίσει. Ήταν πολύ καλή συνεργασία και δεν υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ανδρέας, θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Νομίζω ήταν πολύ καλή η συμφωνία που πέτυχε ο κ. Μπουσόιλ. Αύριο θα περάσει από το Κορεπέρ. Και εφόσον εγκριθεί θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο στη συνεδρία μας, σωστά. Ταχεία διαδικασία λοιπόν. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει συμφωνία, διότι είναι και σφιχτό το χρονοδιάγραμμα. Εάν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο για αυτό το σημείο, θα πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα έως τις 4 που θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα γιατί αυτή την ώρα γνωρίζουν οι συνάδελφοι. Την άλλη φορά έχει προκύψει πρόβλημα για τον ίδιο λόγο, οπότε θα ξαναβρεθούμε στις 4 Να ξεκινήσουμε. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι, λίγη υπομονή, διότι είμαστε στο τελευταίο τριμερή διάλογο για την κοινή αγορά και τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά ως προς την περιαγωγή και την ουδετερότητα του δικτύου, εκεί δεν υπήρξε συμφωνία Οπότε θα περιμένουμε για τη γνωμοδότηση της ΙΜΚΟ σχετικά. Πιστεύετε ότι είναι αρκετοί οι παρόντες για να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ναι. Οπότε να περάσουμε πολύ γρήγορα στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ για όσους ε, δείξατε κατανόηση από σήμερα το πρωί. Θα, μιλήσουμε, θα ψηφίσουμε για την μείωση των ρήπων από τα οχήματα τις οδικές μεταφορές. Ξεκινάμε με την τροπολογία 41 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42-43 υπέρ, κατά, ε, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, ε, εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με την προφορική τροπολογία. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, αποχές, κατά, απόλυτη 47 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 50 υπέρ, όχι, λάθος, είναι συμβαστική 1.51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, 53 υπέρ, κατά, αποχές, which were Απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. I think All right. And you're again, Okay? 12 So 12 against. κατά, 6 υπέρ. Απορρίπτεται. Επόμενη. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, εποχές, απο... Ε, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 και 61 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. 60 και 61. Ίδιο αποτέλεσμα. Α, 12 κατά. 12 προς 7, 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές συγγνώμη δεν έπρεπε καν να την θέσουμε σε ψηφοφορτές πάνω 67 67, 68, 69 unblock υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 70 και 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 12 Πάμε στη 13 τελικά υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ, κατά αποχές. Α, και αυτή έχει καταπέσει. So 75 has fallen. Okay. Πάμε στην τροπολογία 20. Περ. Τροπολογία 20. Σελίδα 8. Πάνω πάνω υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21, 22, 23 και 26 και 29. Αποσύρονται αυτές, άρα θα ψηφίσουμε. Μπορεί να μην το έχετε. Οι τροπολίτες γραπίνη έχουν αποσυρθεί. Τροπολίτες 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται νομίζω να ελέγξουμε. Εγκρίνεται μάλλον, αλλά να ελέγξουμε. Okay. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. λέει 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 26, έχει 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να λέξουμε το 27. Δεν απορρίφθηκε μία, ψήφι, μία ψήφος υπέρ, άρα εγκρίθηκε. Στην τροπολογία 32 πάμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι. Απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 34 κατά 35 και 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 39 δεν την ψηφίζουμε 4 κατά τελική ψηφοφορία ονομαστικά. Plus one. Passed by 20. 20 υπέρ 9 κατά μια αποχή συγχαρητήρια εγκρίνεται.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 θα φτάσει η για το προπολογισμό. Εσεί, Αντρέα θα το αναλάβετε. Α, εντάξει, τέλεια. Υποτίθεται θα μα ενημέρωναν για τη ρομποτική, για τη σχετική του Δεν κατάφερε όμω να είναι εδώ αδελφό. ίσως μετά τον προπολογισμό. Να δώσω στον Αντρέα το λόγο για τον προπολογισμό 2016 την έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα πρέπει να προσέξουμε γιατί θα πρέπει να ακολουθήσουμε λίγο και την ε, σειρά των ε, σημείων της σημερινής διατάξης προκειμένου να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε και στους συντονιστές. Η συνάδελφος Καλτ Σπέλτσε, όπως είπατε, ε, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, δυστυχώς, γιατί έχει καθυστερήσει πτήση της. Γι' αυτό λοιπόν μου ζήτησε να πάρω το λόγο και για το δικό τη το θέμα, το οποίο είναι το θέμα του προπολογισμού και θα το κάνω στα αγγλικά γιατί έλαβα και το σχετικό σημείο μας στα γερμανικά. Η κυρία Καλτσπέρτς μου ανέφερε λοιπόν ότι κατέφεραν, σε ένα δεύτερο σημείο, σε ένα δεύτερο επίπεδο σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του 2016. Γι' αυτό λοιπόν και παρουσιάζει Σήμερα το δεύτερο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τα αριθμητικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει βάσει των στοιχείων αυτών να λάβουμε τις αποφάσεις μας. Το σημείο κίνηση δεν είναι να παρουσιάζει προβλήματα σε ό,τι αφορά τις πιο πολλές γραμμές για την ΕΙΜΚΟ. Ε, καλό αυτό για μας ως Επιτροπή. Οι βασικές προτεραιότητες της προηγούμενου σχεδίου γνωμοδότησης δεν έχουν αλλάξει. Είναι η αγορά, προτεραιότητα αυτό, βασική προτεραιότητα για την πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Και ως εκ τούτου η ομάδα μου συνεχίζει να καλεί για μια έντονη εστίαση σε θέματα διαχείρισης ενιαίας αγοράς ως ένα βασικό θέμα, ένα βασικό ζήτημα ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αλλά εκ παραλλήλου και η προστασία των ε, καταναλωτών θα πρέπει να αποτελεί θέμα προτεραιότητας για να υπάρχει και εμπιστοσύνη από πλευρά των ε, καταναλωτών. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, δημοσιεύσει αποδεκτά αρνητικά στοιχεία για προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχει το θέμα της καταπολέμησης ε, της απάτης και στον ίδιο τον προπολογισμό η κυρία Γκάλπελ θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις και γι' αυτό και καλωσορίζει τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει να στραφούμε και σε ουσιώδη ζητήματα. Καταρχάς, ε, τα μέτρα που υπήρχαν ήδη για το φόρουμ της ενιαίας αγοράς. Η συγκεντρία πιστεύει ότι στο θέμα αυτό, από δική μας πλευράς, θα μας βρει ενωμένου όλοι αν αναγνωρίζουμε ε, πόσο σημαντική είναι η συνέχιση της χρηματοδότησης του ετησίου φόρουμ που ε, χρηματοδοτείται από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου. Αλλά προφανές η Επιτροπή είναι αυτή που διοργανώνει την εκδήλωση. Και θέλουμε να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η εκδήλωση αυτή, γιατί έρχονται σε επαφή οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις ε, για να επιδείξουν την δασμευσή τους για την ε, εφαρμογή τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά. Η συγγήτριά μα λοιπόν μα επιθυμίζει επίση ότι πρόκειται ότι τελευταίο έτο ε, προπαρασκευαστικό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανώσει την συνέχεια του γεγονότο αυτού για να διασφαλίσει τη σημασία του στην ενιαία αγορά. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, η δική μα Επιτροπή έκανε μια σύσταση για τη χρηματοδότηση ενό νέου πιλωτικού προγράμματο για τον καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή. Και έτσι λοιπόν θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις και να, να εξηγήσουμε τις ε, προκλήσεις που συνδέονται με, την, ε, με το εμπόριο. Αυτά θα τα αποφασίσουμε βέβαια και μετά από διαβούλευση με τους συναδέλφους. Επειδή δεν έχουμε τόσε πολλέ πληροφορίε. Θα θέλαμε να καλέσουμε του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μα παρουσιάσουν στην Επιτροπή πώ έχει τρέχουσα κατάσταση. Και τα άλλα, κυρία Πρόεδρε, η σκιώδη εισηγήτρια ζητά από την Κριστίνη Σφέμπερ για τα πρακτικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά τα θέματα του Single Market Forum να μας αναφέρουν κάποια στοιχεία τα οποία θα είναι χρήσιμα για την σκιώδη ηγετρία. Αυτά λοιπόν έχει να παραθέσει η σκιώδη ηγετρία και ευχαρίστω να ακούσουμε τα σχόλια των συναδέλφων και θα τα αναφέρω. Ευχαριστώ. Τώρα στράφουμε προ το σκιώδη, λέει η πρόεδρο. Δεν βλέπω εδώ τον σκιώδη από τον. Ε, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η Εύελιν θα πάρει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της κυρίας Γκαλπίνη, η οποία δεν μπορεί να έρθει στις Βρυξέλλες αυτήν την εβδομάδα. Έχει μεγάλες υποχρεώσεις στην πατρίδα της ε, και γι' αυτό λοιπόν μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω εδώ σήμερα. Μας ενημερώνει λοιπόν ότι είναι ευγνώμων για την πολύ καλή συνεργασία με την εισηγήτρια την κυρία Καλπέλτς η οποία επέδειξε πολύ ανοιχτό πνεύμα όντως. Αυτά λοιπόν τα οποία παρουσιάζει ως προτάσεις η κυρία Καλπέλς αποτελούν μια εξαιρετική βάση και αποτελούν και μια συνολική πρόταση βάση της οποίας θα συνεργαστούμε πολύ καλά. Κάποιους από τους τομείς αυτούς θεωρώ ότι τους ανέφερε ήδη ο συνάδελφος ΣΒΑΠ, η κυρία Γκραπίνη θα ήθελε άλλη μια φορά να θέσει στο επίκεντρο το θέμα της γραμμής προϋπολογισμού με ένα νεοποιητικό πρόγραμμα για την ψηφιακή αγορά. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα και μια καλή συνέχεια σε αυτά που συμφωνηθήκαν το 2015 σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση για την ψηφιακή εποχή για την ε, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ χρήσιμο θεωρώ και θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να το προσεγγίσουμε. Η κυρία Κραπίνη θεωρεί επίσης ότι δεν έχει σχεδόν τίποτε να προσθέσει στο κείμενο μόνο κάποιες μικρές λεπτομέρειες θα εισαγάγει, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν σε καμία περίπτωση την πρόταση της κυρίας Γκαλπέλτς. Πρόκειται για κάποιες μικρές προσθήκες ε, ή διευκρινήσεις αν θέλετε. Κατά τα άλλα όμως, εμείς ως σοσιαλδημοκράτες είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε πλέον μπροστά μας. Σας ευχαριστώ. και τώρα να στραφούμε προς τον σκιάβε του ECR των συντηρητικών των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Την Κρυτάλτον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τη δική μας την Σκοπιά, γενικώ η πρόταση είναι καλή. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά του εισαγητού Αλλά έχω παρόλα αυτά ένα σοβαρό δίλημα. Διότι τη δική μας την ομάδα, γενικώς από την... Η αρχική μας θέση είναι να μην δεχόμαστε περισσότερα πιλωτικά προγράμματα για περισσότερες προκύπασεις όσο ήδη ισχύουν. Όμως, πρόταση του συγητή, όσο καλή κι αν είναι, και όσο και σε κάποια ζητήματα δείχνει στήριξη στην πραγματική οικονομία, την μικρομεσαίε, την δημιουργία θέσεων απασχόληση για την τόνωση τη οικονομία, και αυτά μπορούμε να τα στηρίξουμε. Πιστεύουμε ότι παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχουν περισσότερα χρήματα, περισσότερα κονδύλια για τα μέτρα εσωτερική αγορά. Εκεί χρειάζεται καλύτερη επιβολή των μέτρων. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξουν εξοικονομήσει από άλλα τμήματα του προπολογισμού. Δυστυχώ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί έχει άλλου τομεί προτεραιότητε η Επιτροπή. Αλλά κατά τα άλλα στηρίζουμε τη γνωμοδότηση αυτή και θα συνεργαστούμε επικοδομητικά για να κάνουμε καλέ προτάσει σε άλλου όμω τομεί του προπολογισμού, διότι στον κοινωνικό προπολογισμό συνολικά πρέπει να δούμε πού ε, μπορούν να γίνουν εξοικονομήσει για να δαπανηθούν περισσότερα κονδύλια για τα μέτρα εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα από του φιλελευθέρου η Δίτα. Ευχαριστώ. Θα επαναλάβω αυτό που είχα πει και τον περασμένο μία, μήνα, ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την γνωμοδότηση. Συμφωνώ και θα υποβάλω τροπολογίες και για την προηγούμενη γνωμοδότηση. Όσο για τα πιλωτικά προγράμματα και η δική μας ομάδα συμφωνεί και θα ενημερώσουμε του συναδέλφου Επιτροπή Προπολογισμών να στηρίξουν και αυτοί στι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό και για το ε, συνολικό πακέτο. Ευχαριστούμε, Ντίτα. Δεν έχω άλλα ονόματα από τους σκιώδεις. Δεν ξέρω αν η Πράσινη, η Γκουε ή η FDD έχει κάτι να πει, έχουν κάτι να πούν. Συνάδελφοι, Ρόζα, Ρόζα παρακαλώ. Thank you um, ευχαριστώ πολύ. Η συνεργασία με την κυρία Γκάλι Πέλτσα ήταν μόνο ταξί της ιδέας και των σκιωδών, αλλά και με τους υπολείπους. Σε ό,τι αφορά αυτή τη γνωμοδότηση για τον προπολογισμό. Δύο σημεία που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα θέλω να αναφέρω. Το πρώτο. Είμαι γνώμων να υπάρξουν χρήματα για το ODR, την επίσημη αντιξιακή βοήθεια. Κάτι γίνεται ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βρεθούν πόροι. Ε, πρέπει να επαγρυπνούμε και εμείς. Σε ό,τι αφορά δε την ενιαία αγορά. Παρακαλώ όλοι να συμμετέχετε από νωρί προετοιμασίες για να μην τα κάνει μόνη τη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίτερα για την μια αγορά στον τομέα των ψηφιακών, της ψηφιακή τεχνολογία επίση. Για την εκπαίδευση, δασκαλία, κατάρτιση, το 7ο σημείο. Το φόρουμ της αγοράς. Πρέπει να ασκήσει κάποια πίεση. Η ίδια εκδήλωση έχει ως στόχο την πληροφόρηση και είναι ένα ενημερωτικό εργαλείο ή εκδήλωση, όπως θέλετε πείτε προώθηση προώθησης, προβολής και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο. Τέλος. Δεν θα έπρεπε. Θα το σκεφτούμε κι εμείς. Ε, και εγώ προσωπικά όταν θα έρθει η ώρα να καταθέσουμε τροπολογίες μήπω θα έπρεπε, λέω, για την πληροφόρηση και για την πρόθεση τη ένα αγορά. Μήπω θα έπρεπε να ε, χρηματοδοτήσουμε την ερωτική εκστρατεία, γιατί οι πολίτε δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα. Έχουμε το Solvit στον προπολογισμό, για παράδειγμα, αλλά έχουμε πολύ και πάντα είχαμε πολύ λίγα χρήματα για την πρόθεση του Solvit. Άρα ελάχιστοι είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες που χρησιμοποιούν τα εργαλεία που υπάρχουν στην ενιαγορά αγορά ή τις ενημερωτικές τα κτλ. Ελπίζω λοιπόν να είναι αυτό μια καλή ευκαιρία για να επιστήσουμε την προσοχή της κοινής γνώμης. Ευχαριστώ τη Ρόζα. Στρέφομαι προς άλλους συναδέλφους, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Δεν βλέπω κάποιον άλλο. Νομίζω έχουμε κάποιους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αίθουσα. Η Κομισιόν λοιπόν, παρακαλώ. Ήρθε και η συγγήτρια όμως. Να καθίσει πρώτα η συγκεκριά μας. Πολύ γρήγορα ήρθε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της συναδέλφου, η οποία κρατάνει όπου να είναι. Νομίζω ότι είμαι στην εξαιρετική κατάσταση και σε μοναδική θέση να μπορώ να σα κάνω αρκετά χαρούμενους, γιατί σε ό,τι αφορά το Single Market Forum θα προσπαθήσουμε με την εβδομάδα των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων να τα συνενώσουμε τα δύο έργα αυτά και έτσι να εξυπηρετήσουμε την συζήτηση και την εναρμόνιση και την ενημέρωση και να βρούμε και τη θετική ενέργεια που χρειάζεται. Αυτό σημαίνει από πλευρά χρηματοδότηση θα πρέπει να βρούμε τη σχετική ενέργεια και επιφωλάσσομαι για την οριστική απόφαση, αλλά δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει η ανάγκη να ψάξουμε να βρούμε νέα νομική βάση, γιατί τα εφιστάμενα μέσα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, μπορούμε να, επεν... να... να εγγυηθούμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει στην παρούσα μορφή το Single Market Forum, αλλά θα ενσωματωθεί πιο πολύ με, τη μικρομεσαία, με τις της μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χωρίς να σας κουράσω μόλι λεπτομέρειες. Αυτό ήταν η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν αυτά είχα να σας αναφέρω στο διαφορά του Single Market Forum. Thank you. I'm just going to hand to our rapporteur to give her a few moments. Η συγγήτρια. Ελπίζω να μην ε, λαχανιάσετε μέχρι να φτάσετε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη που άργησα. Αλλά είχε πάνω από μια ώρα καθυστέρηση πτήση μου Θέλω να ευχαριστήσω πάντως όλους όσους με βοήθησαν να, ε, να καταρτήσω την νομοδότηση αυτή. Νομίζω ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Από κοινού επεξεργαστήκαμε την πρόταση και πρόκειται για μια κοινή πλέον θέση. Βέβαια, αυτό που είπε η Κομισιόν με λυπεί κάπως. Ότι δηλαδή τα μέτρα σε αφορά το φόρουμ της ενέας αγοράς δεν θα συνεχιστούν όπως τουλάχιστον εμείς θα επιθυμούσαμε. Θα δούμε βέβαια πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τα σχετικά στα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να ιεραρχήσουμε σωστά τις προτεραιότητές μας. Γιατί και τα δύο μέτρα είναι εξίσου σημαντικά. Και έχει νόημα και σημασία και η προοπτική που θα τους δώσουμε. Δεν είναι μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι καταναλωτές ή και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αυτό το φόρουμ της εννέας αγοράς και οι καταληκτικές μας παρατηρήσεις στην έκθεση θα πρέπει να είναι ισορροπημένες, θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση και στο μέλλον για να μην χαθεί τίποτα από αυτές τις μέτρων καλό θα ήταν ίσω να τα προτείνουμε στο πλαίσιο μιας νέας νομοθετικής πρόταση. Λυπούμε και πάλι που καθυστέρησε και σα ευχαριστώ για τη βοήθεια και τη συνεργασία. Πρόεδρο, θέλει η Κομισιόν ξανά το λόγο, Ενδεχομένω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως ε, να μην εκφράστηκα αρκετά με σαφήνεια. Το Single Market Forum θα συνεχίσει να υφίσταται. Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε θέματα ε, ε, χρηματοδότηση, μάλλον θέλουμε να συνενώσουμε από πλευράς περιεχομένου και χρηματοδότηση με την εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν είναι φυσικά όλα τα θέματα του φόρουμ, δεν άπτονται όλα τα θέματα του φόρουμ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχει δίκιο λοιπόν η συγγεντρία, ούτε προ, προτιθέμεθα να κάνουμε αυτό. Όχι, αναζητούμε μια συνεργασία και χρηματοδοτική αλλά και από πλευρά περιεχομένου προκειμένου να προωθήσουμε την κατάσταση αυτή. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση το Single Market Forum να σταματήσει. Αυτό για να μην υπάρξει παρανόηση. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, σας ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Παρακαλούμε κυρία Γκέπχαρτ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω μια παρατηρήση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την διευκρίνηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω το εξή. Αυτή η ιδέα του Φόρουμ Εσωτερική Αγορά ε, ήρθε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιλαμβάνονταν και σε μία έκθεση τη συναδέλφου του Χουνστάιντ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρόζα, για την εξαιρετική αυτή ιδέα. Αλλά θα ήταν πάρα πολύ καλό αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έπαιρνε πάνω της όλη την προετοιμασία, αλλά αν θα μπορούσε να συμπεριλάβει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην φάση της προετοιμασίας, προκειμένου να μπορούμε να αποστείλουμε όχι μόνο ένα-δυο άτομα να παρακολουθούν, αλλά να είμαστε και στην, στο μέλλον ένα μέλος του φόρουμ, ένα πραγματικό μέλλον και ε, μέλος του φόρουμ αυτού. Και νομίζω ότι η Ρόζα συμφωνεί μαζί μου και τουλάχιστον να γνέψει καταφατικά. Ευχαριστώ. Για πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Καταφτάσατε μόλις βέβαια. Έχουμε προχωρήσει και πιο πολύ από ό,τι προβλεπόταν στην ημερήσια διάταξη. Δεν θέλετε να πάρετε το λόγο. Έχουμε, έχουμε λίγο χρόνο. Με συγχωρείτε, αλλά τα πάντα είναι μπλοκαρισμένα έξω από το κοινοβούλιο, υπάρχει περιορισμένη κυκλοφορία. Εγώ χρειάστηκε να σταθμεύσω μακριά. Ναι, ναι, όλοι τα γνωρίζουμε αυτά εάν θέλετε να πάρετε το λόγο παρόλα Ναι. Ήδη μιλήσαμε για τη γραμμή του προπολογισμού που αφορά αυτά τα θέματα. Όπως ήδη εξήγησε ο συνάδελφος, μας απασχολούν όλες οι διαφορετικές επιλογές. Όμως τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει με την συγχώνευση της νέας γενικής διεύθυνσης για την αγορά με αυτή των επιχειρήσεων. Έχουμε νέες δυνατότητες λοιπόν, κοιτάζουμε όλες τις επιλογές αλλά ίσως να βρούμε άλλους τρόπους να διασφαλίσουμε το φόρουμ για την εσωτερική αγορά. Σας το λέω γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό και θεωρούμε ότι είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα σε τόσο δύσκολους καιρούς και μπαίνοντα κατάλαβα ότι όπως είπε και η κυρία Γκέμπχαρτ το Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως στην ανανέωση του φόρουμ της ενίας αγοράς. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Είχαμε ανταλλαγέ με κάποιου από του ευρωβουλευτέ και από διαφορετικέ ομάδε και καλωσορίζω όλε αυτέ τι ιδέε. Θα έχουμε συγκεκριμένα εργαστήρια και του χρόνου ένα μεγάλη σημασία γεγονό επί Ολλανδική Προεδρία. Με συμμετοχή διαφορετικών ομάδων και επιμέρου βουλευτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το θέμα. Θα ακούσατε εδώ ότι στηρίζουμε το φόρουμ τους, ε, της ενιαίας αγοράς. Μιλήσατε για δυνατότητα συνεργασία στο μέλλον ε, και εμείς θέλουμε να ενημερωνόμαστε για όσα γίνονται και σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Αυτή είναι η πρώτη μας συζήτηση, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 14 Ιουλίου το μεσημέρι. Εξέταση των τροπολογιών στις 30 Σεπτεμβρίου ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ στις 3 Σεπτεμβρίου. Θα παραμείνουμε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα λοιπόν και μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση για αυτό το σημείο. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίασής μας. Υπάρχουν διάφορα που θα ήθελα να συζητήσουμε οι συνάδελφοι. Όχι, οπότε συνάδελφοι να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 15 Ιουλίου στις 9 και θα σας καλωσορίσω εκεί. Σας ευχαριστώ. Κυρίζω τη λήξη.